przewodniczący! Please take your seats. Καθίστε παρακαλώ, συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος. It's just three minutes past three. Τρία, τρεις και τρία. Είναι λέει ο πρόεδρος, γιατί πάει λάθος το ρολόι, πάει πίσω, άρα πρέπει να αρχίσουμε. Παραφτήκα. Στα πολωνικά. Συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Είχαν σταματήσει 21η Δεκάτου του ενεστώτος έτους. Τα οι ποσεδενια 21 Τα πρακτικά τη συνεδρίαση τη 21 η Δεκάτου διατίθενται και σας ρωτώ για έχετε κάποιες παρατηρήσεις. Δεν βλέπω καμία ένσταση, επομένως εγκρίνονται τα πρακτικά εκείνα. Και θα προβάλλω τώρα εις κάποιες ανακοινώσει. Πώς δεν λειτουργεί η μετάφραση, η διερμηνία. Λέει τρεις φορές ο πρόεδρος. Now it's okay. Α, τώρα δουλεύει. Σας ρώτησα για τα πρακτικά της 21ης Οκτωβρίου. Μήπως έχετε παρατηρήσεις. We accepted the minutes. Αφού δεν έχουμε ενστάσεις, θεωρούνται εγκεκριμένα. Πριν αρχίσει η συζήτηση θα πρέπει να σας πω ότι στις 6 Νοεμβρίου ο Ολέγκ Κάσιν υπέστη επίθεση και ξυλοδαρμό. Πρόκειται για πράξη που θα πρέπει να καταδικαστεί. Θεωρούμε πάρα πολύ θετική την ταχύ αντίδραση των ρωσικών αρχών και το ότι ο πρόεδρος Μέντβεντεφ προσωπικά ασχολήθηκε με την σύλληψη των Υπετίων. Στις 21 ε, Οκτωβρίου, για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, έγινε διαδήλωση της αντιπολίτευσης στην κεντρική πλατεία της Μόσχας. Θεωρούμε ότι πρόκειται για θετικό γεγονός και αντιστοίχως και εμείς έχουμε ζητήσει περαιτέρω δημοκρατισμό της χώρας και επομένως βλέπουμε ότι οι ενέργειές μας έχουν πιάσει τόπο. Τρίτον, πριν από κάποιες μέρες στην Βαγδάτη ε, σημειώθηκε επίθεση κατά χριστιανών οι οποίοι ασκούσαν τη λατρεία τους σε κάποια εκκλησία είχαμε θανάτους αλλά και τραυματίες για άλλη μια φορά θα πρέπει να απευθύνουμε έκκληση προς πάντες να σεβαστούν την ε, ελευθερία της ε, θρησκευτικής λατρείας και ότι θα πρέπει να καταδικαστεί κάθε βία ενέργεια τέταρτον στις 10 Δεκεμβρίου πρόκειται να λάβει μια χώρα, ούτω, χώρα μια εκδήλωση για την απονομή του βραβείου Νόμπελ. Οι δε κινέζικες αρχές έχουν προσπαθήσει να πιέσουν τα κράτη-μέλη να μην γίνει η εκδήλωση αυτή. Εμείς πάντως ε, πρεσβεύουμε το να τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα παντού και στην Κίνα. Κατά την εκδήλωση εκείνη θα εκπροσωπηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον επικεφαλή τη εκείνη την προσωπία τη Ένωση. Έχουμε τώρα κάτι διαδικαστικού χαρακτήρα. Θέλω τον λόγο κύριο Μπέλιγκερ. Τι φυσικέ καταστροφέ φοβερή ε, ε, ένταση χτύπησαν την περιοχή τη Ιταλία στο Βένετο πρόσφατα, Βιτσέντσα, Πάντοβα και Βερόνο. Ε, πρόκειται περί πλημμυρών καταστροφικών διαστάσεων που δημιούργησαν οι βροχοπτώσει περίπου 500.000 500 άτομα που επλήγησαν αυτόν τον τρόπο και εκατοντάδε χιλιάδε ευρώ σε ζημιέ. Ε, τραγωδία γονάτισε όλε τι παραγωγικέ περιοχέ, τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και διάφορου τομεί. Απευθύνω έκκληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στου συναδέλφου, ούτω ώστε στα όρια των οργανισμών προβλέπουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύη και τα Διευθυντικά Ταμεία, στα όρια αυτά να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για να υποστηριχθούν αυτοί οι πληθυσμοί και να βρεθούν κάποιε λύσει για να βρεθεί μια απάντηση σε τέτοιε καταστροφέ. Να να πω, να πω και κάτι άλλο διαφορετικό, ότι η Ιταλία, η χώρα μας, σήμερα έχει κι άλλο λόγο για να θρυνεί καταστρεφεί, ε, καταραίει πομπία. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό δυστυχώς το γεγονός και χρειάζεται να ρίξει μια ματιά και σε τέτοια πράγματα η Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Και επίσης παρακαλώ να αναφερθείτε σε αυτό